Hello everyone, if you can take your seats, we can start the meeting. First of all, if you agree with agenda, then... Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Αν συμφωνείτε λοιπόν, θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, ως συνήθως η συνεδρίασή μας μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Έχουμε διευμηνία σε 22 γλώσσες. Έχετε τις αποφάσεις των συντονιστών της 25ης Σεπτεμβρίου στο φάκελό σας. Να σας πω τι έγινε με τον προϋπολογισμό και την ε, στροπολογίες για τον προϋπολογισμό που κατατέθηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου. Εμείς είχαμε ζητήσει αυξήσεις για στρατηγικού ενδιαφέροντος γραμμές Εν τω μεταξύ η Επιτροπή Προϋπολογισμών ψήφισε την 1η Οκτωβρίου όλες τις τροπολογίες που είχε δεκτεί και σύνεπως το αποτέλεσμα για την Ήτρε είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό με σημαντικές αυξήσεις για την έρευνα, για τις μικρομεσαίες, για το διάστημα και για άλλους τομείς τους οποίους είμαστε υπεύθυνοι. Ελπίζουμε ότι η Ολομέλεια λοιπόν θα ακολουθήσει την ίδια γραμμή την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε ένα εξαιρετικό πακέτο για τις διαπραγματεύσεις από πλευρά του Κοινοβουλίου. Και ευχαριστώ όλα τα μέλη τα οποία πήραν μέρος σε αυτή την προσπάθεια και ελπίζω και τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν ότι ένας τέτοιος προπολογισμό για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι κάτι το προαπαιτούμενο για το 2020. Σύμφωνα τώρα με το άρθρο 241 οι νομομαθείς των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου προετοίμασαν ε, μια πρόταση για τις στατιστικές των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει διανεμηθεί το κείμενο σε όλες τις γλώσσες στις αρχές Οκτωβρίου με ένα διορθωτικό. Λόγω του περιορισμού ε, του χρονικού δεν υπήρχε γλωσσικός έλεγχος και αναθεώρηση των κειμένων. Η διαδικασία για την υιοθέτηση τώρα αυτού του διορθωτικού είναι η εξής. Τη απουσία ή ασδήποτε αντιρρήσεως μετά από την ανακοίνωση που έκανα τώρα, το διορθωτικό θα υποβληθεί απευθείας στην Ολομέλεια στις 21 Οκτωβρίου και θα πρέπει να υποστηριχθεί από 38 μέλη τουλάχιστον ε, Λοιπόν, δεν έχω κάποιες άλλες παρατηρήσεις τώρα να κάνω, ανακοινώσεις, συγγνώμη. Ε, πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου. μέχρι το τέλος του χρόνου, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα θεωρηθούν δεκτά. Να καλωσορίσω τώρα τον κύριο Μπόκθατ, ε, αναπληρωτή διευθυντή της GNR στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα έχουμε μαζί του σήμερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία των κατεξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με τα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος, PCI, διαμεθοριακά προγράμματα, ενεργειακά συστήματα, διανομή ηλεκτρισμού. Θα θα βοηθήσουν να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργειακή της πολιτική και τους στόχους στον τομέα των περιβάλλον, του περιβάλλοντος στις μεθοριακές περιοχές και στους λεγόμενους θυλάκους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε δύο χρόνια καταρτίζει ένα, ένα νέο ε, πρόγραμμα τέτοιου είδους κοινού ενδιαφέροντος προγρα, ε, κατάλογο. Έχουμε καλέσει λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει και το ποιες θα είναι η κατεξουσιοδότηση πράξης γύρω από τα PCI στο μέλλον. Να θυμίσω ότι ε, όταν υιοθετήσει μια κατεξουσιοδότηση πράξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί για έλεγχο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έχουμε την δυνατότητα να την εξετάσουμε για ένα δίμηνο, έχουμε δυνατότητα να αιτηθούμε παρατάσεως για άλλο ένα μήνα και στο τέλος να εγκρίνουμε την πρόταση ή μη. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα για την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε που μας στείλατε ήδη από χθες τον κατάλογο και θα ακούσουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας κάνετε κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις <coughs> σχετικά με τον κατάλογο αυτό, όπως επίσης και κάποια σχόλια για το χρονοδιάγραμμα έγκρισης αυτού του καταλόγου. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. για τον κατάλογο των προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όπως ακούσατε ήδη χθες το απόγευμα. Σας στείλαμε τα απαιτούμενα έγγραφα. Δεν θα υπάρξει συζήτηση σε βάθος, ε, αλλά ε, σε κάποια άλλη φάση θα μπορέσουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω σε αυτή την εισαγωγική φάση είναι να σας δώσω μια ιδέα της σημασίας και των αποτελεσμάτων των διαδικασιών που οδήγησαν μέχρι τώρα σε, σε αυτή την πρόταση του καταλόγου των προγραμμάτων. Και φυσικά να έχουμε και λίγο χρόνο για ανταλλαγή απόψεων. Ας ξεκινήσω λοιπόν με κάποιες διαφάνειες. Εδώ υπογραμμίζω την σημασία που έχει ο κατάλογος PCI και για τα ενεργειακά συστήματα τα οποία συνδέονται με τις υποδομές Αυτός είναι ένας κλάδος, αν θέλετε, ένας τομέας ο οποίος αλλάζει συνεχώς και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να, να είναι σε μόνιμη υποεξέταση. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω εδώ είναι η σημασία που έχουν οι υποδομές. Οι υποδομές θα πρέπει να υπηρετούν στην ουσία και τους τρεις στόχους της ενεργειακής μας πολιτικής, δηλαδή αηφορία από τη μία, οι υποδομές θα πρέπει να υπηρετούν λοιπόν και τις προσπάθειες ανάπτυξη ε, και αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να βοηθά στην διασφάλιση της προμήθειας ενέργειας. Να έχουμε τις σωστές υποδομές σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα οι χώρες ε, να τους παρέχεται εν πάση περιπτώσει η ενέργεια η οποία χρειάζεται για ηλεκτρισμό, για θέρμανση, ε, ψήξη κτλ. Και τρίτον είναι η ανταγωνιστικότητα και η διαθεσιμότητα. Προφανές είναι ότι μπορεί κανείς να φανταστεί ένα τέλειο δίκτυο με υψηλό κόστος αλλά κάποιος θα πρέπει να τα πληρώσει όλα αυτά. Και γι' αυτό ακριβώς γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός, είναι ο τελικός χρήστης, είναι ο καταναλωτής. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε όταν αναπτύσσουμε κάποια δίκτυα υποδομών να επιλέγουμε τις δυνατότητες οι οποίες έχουν το μικρότερο δυνατό και αποδοτικότερο κόστος. Τώρα γιατί υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον συμπερίληψη στον κατάλογο PCI. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο κανονισμός προβλέπει ότι το PCI θα πρέπει να συνοδεύεται από μια διαδικασία διοδότησης επιταχυμένη και ταυτόχρονα όλες ε, ακριβώς αυτές οι χορηγήσεις αδειών θα πρέπει να περνούν ε, μέσω ενός one-stop shop. Έχουν ένα ειδικό λοιπόν διακανονιστικό πλαίσιο τα PCI, κάτι το οποίο διευκολύνει την εφαρμογή τους. Παράδειγμα, ε, μία από τις προϋποθέσεις για τις χώρες στις οποίες θα εγκατασταθούν αυτά τα προγράμματα, δύο τουλάχιστον, θα πρέπει να αποδέχονται τις προτάσεις αυτές εκ των προτέρων έτσι ώστε να μην υπάρχουν επιφυλάξεις εκ των υστέρων σε πολιτικό ή οικονομικό επίπεδο. Είναι μια επιπλέον εγγύηση για τα PCI. Και τρίτον, και εδώ είναι το πιο σημαντικό για τους υπεύθυνου, είναι η οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε μία άμεση διασύνδεση ανάμεσα στα PCI και στα Connecting Europe. Μπορούμε να αποδεχθούμε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης στα πλαίσια του Connecting Europe εφόσον εκ των προτέρων έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των PCI. Για να καταλάβετε λίγο περισσότερο αυτά τα οποία έχετε κάνει και έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, να πω ότι στα πλαίσια αυτού του κανονισμού Έχουμε χρηματοδοτήσει και μελέτες και προγράμματα, 67 δράσεις στον τομέα του ηλεκτρισμού, 2,1 δις, 65 δράσεις στο φυσικό αέριο, 1,5 δις, 4 δράσεις στα λεγόμενα ΕΦΗ e δίκτυα, 134 εκατομμύρια και 3 δράσεις για το διοξίδιο του άνθρακα, 9,7 εκατομμύρια. Πρόκειται για μια προκαταρκτική αξιολόγηση γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε ακόμα ένα χρόνο, ο επόμενος χρόνος είναι ε, ο τελευταίος του πρώτου συνόλου προγραμμάτων. Το επόμενο θέμα είναι στην ουσία ε, μια περιγραφή της διαδικασίας. Πώς επιλέγονται τα προγράμματα αυτά, τα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος, PCI. Ο χώρος για την ανάπτυξη των PCI ε, θα έλεγα ορίζεται από τις περιφερειακές οντότητες. Οι ομάδες οι περιφερειακές, οι ομαδοποιήσεις οι περιφερειακές ε, καθορίζουν τη μεθοδολογία. Σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό, για να σας δώσω ένα παράδειγμα σε σχέση με τον κανονισμό 10E, σχετικά με τα κριτήρια επιλογής ενός προγράμματος, ένταξη στην αγορά, βελτίωση ανταγωνισμού, διασφάλιση προμήθειας και αηφορία. Αυτά είναι τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση της λεγόμενης πλατφόρμας συνεργασίας. Οι περιφερειακές ομάδες προετοιμάζουν λοιπόν έναν κατάλογο μετά από μακρόχρονες συζητήσει και ο κατάλογος αυτός προτάσεων ε, καταλήγει στο σώμα το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις. Σε επίπεδο περιφερειακής ομάδας υπάρχουν και τα λεγόμενα critical projects. Τα κρίσιμα προγράμματα. Ναι, μεν υπάρχει, ε, υπάρχει η απλή λογική που κυριαρχεί στον τομέα, η κοινή λογική στον τομέα της κατάρτισης των προγραμμάτων, αλλά πολλές φορές ε, υπάρχει μια, θα έλεγα, η ιδιαίτερη υπογράμμιση συγκεκριμένων προγραμμάτων για άλλους λόγους, όχι για αυτούς που προβλέπονται. Ως εκ τούτου αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να συζητιώνται ακόμα περισσότερο και οι περιφερειακές ομάδες είναι αυτές που αποφασίζουν το τι θα υποβληθεί στο σώμα λήψης αποφάσεων. Οι ομάδες λήψης αποφάσεων είναι οι ομάδες που αποτελούνται, που συνίστανται από τους γενικούς διευθυντές των αντίστοιχων Υπουργείων των κρατών μελών. Η περιφερειακή αυτή ομάδα θα πρέπει με συνένεση να παίρνει αποφάσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί όπως σας είπα ήδη υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν ε, ξεκάθαρο πολιτικό περιεχόμενο για κάποια κράτη-μέλη, θα μπορούσαν να υπάρχουν, δεν έχει συμβεί αυτό. Θεωρητικά λοιπόν θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο κρίσιμο πρόγραμμα, το οποίο είναι αμφισβητήσιμο, να οδηγήσει στο μπλοκάρισμα του συνόλου της διαδικασίας και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει κανείς έξω από μια τέτοια διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα πιο σύγχρονο τρόπο επιλογής στα πλαίσια αυτά. Εγώ είπα ότι μέχρι πριν δύο εβδομάδες ε, ε, έγινε μια συνεδρίαση αυτής της ομάδας λήψης απόφασης και υπήρξε συνένεση για όλα τα προγράμματα, οπότε το θέμα τίθεται σε θεωρητική προς το παρόν βάση. Τώρα, ε, για τον χρονισμό δεν ξέρω, ε, μπορεί κανείς να θέλει να περάσει σε λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής από την πλατφόρμα συνεργασίας, στην περιφερειακή ομάδα, στην ομάδα λήψης απόφασης, έχουμε θα έλεγα μια ανοιχτή διαδικασία, μια ξεκάθαρη διαδικασία. Έχουμε πολλαπλές ε, συναντήσεις, ε, έχουμε συναντήσεις με web streaming, Έχουμε πολλαπλές διαβουλεύσεις και από πλευρά ε, του τρίτου καταλόγου, της τελευταίας συζήτησης που κάναμε, έχουμε μια εντατική συμμετοχή των μελών του ιδίου του κοινοβουλίου σας. Και φυσικά περιμένουμε με αδημονία τα σχόλιά σας. Έρχομαι τώρα στα βασικά στοιχεία του τέταρτου καταλόγου σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος. Βλέπετε ε, κάποιες εξελίξεις σχέση με τον προηγούμενο, τον τρίτο κατάλογο σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος. Το πρώτο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι έχουμε μείωση των σχεδίων κατά 30%. Από 173 έχουμε 151 σχέδια. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά επιμείναμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο γεγονός ότι όλα τα σχέδια που δεν σημείωσαν πρόοδο ή σημείωσαν ανεπαίσθητη πρόοδο τα τελευταία δύο-τέσσερα χρόνια να αφαιρεθούν από τον κατάλογο. Γιατί η έλλειψη πρόοδου είναι ένδειξη ότι υπάρχει πρόβλημα με την δρομολόγηση του σχεδίου. Οπότε η αφαίρεσή του από το σχέδιο του καταλόγου δεν σημαίνει ότι έχει καταδικαστεί ε, για πάντα. Μπορεί να επανέλθει όταν έχει οριμάσει η πορεία του. Αλλά Σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν να μην έχουμε ένα πληθωριστικό αριθμό σχεδίων όταν γνωρίζουμε ότι μερικά από αυτά στην επόμενη διετία δεν πρόκειται να αναπτυχθούν δεόντως. Γι' αυτό τα αφαιρούμε. Έτσι λοιπόν εξηγείται αυτή η μείωση του αριθμού των σχέδιων. Τώρα, πώς εντάσσεται αυτή η μείωση στα διάφορα σχέδια ενεργειακών υποδομών. Έχουμε μία μικρή μείωση στα σχέδια του ηλεκτρισμού, 4%. Έχουμε μεγάλο αριθμό σχεδίων φυσικού αερίου που αφαιρέθηκαν, 40%. Επίσης έχουμε αύξηση των σχεδίων έξυπνων δικτύων, ήταν όμως ήδη σε πολύ χαμηλά επίπεδα, οπότε έχουμε 15% αύξηση, αλλά αν έχουμε από, αύξηση από 2 σε 4 σχέδια δεν είναι πολλά. Και επίσης 25% για τα δίκτυα διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα, να δούμε τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δικτύων. Ενέργειας, ηλεκτρισμού μάλλον, έξυπνο δικτύο κτλ. Από την αρχή είπαμε, μια και υποστήριξαμε τα σχέδια φυσικού αερίου, το είχαμε πει από την αρχή ότι λόγω της οριμότητας πολλών τέτοιων σχεδίων θα έχουμε πολύ περισσότερα σχέδια φυσικού αερίου στην αρχή του συστήματος Στη συνέχεια όμως θα υπερκεραστούν από τα σχέδια του ηλεκτρισμού, κάτι που έχει αποδειχθεί στον τέταρτο κατάλογο. Εδώ στον τρίτο κατάλογο είχαμε δύο προς 1 την αναλογία, στον τέταρτο κατάλογο έχουμε τρία προς 1. Και πιστεύουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Αυτά εν είδη εισαγωγής. Θα ήθελα λοιπόν τον υπόλοιπο χρόνο να τον αξιοποιήσουμε για ανταλλαγή απόψεων και περιμένω με ανυπομονησία τις ερωτήσεις σας και τις, ε, τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Πόρτσαρτ. Θα έχουμε πρώτα ένα γύρο με τους συντονιστές και φυσικά όποιος συνάδελφος επιθυμεί στη συνέχεια να λάβει το λόγο να το δηλώσει στη γραμματεία. Η κυρία Καρβάλιο. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και το καλεσμένο μας για την παρουσίαση του σχεδίου του τετάρτου καταλόγου των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος. Δεν φαίνονται καλά οι διαφάνειες από εδώ, κυρίως ε, προς τα αριθμητικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαφάνεια σε σχέση με την προηγούμενη, δεν ξέρω αν υπάρχει και σε χαρτί. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζω ότι δυστυχώς ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή είναι πολύ περιορισμένος. Πάντως θα θέλαμε πολύ περισσότερη ανάμιξη και καλύτερη ενημέρωση της όλης διαδικασίας. Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερος. Δεύτερο σχόλιο. Κατανομή των σχεδίων. Στην προηγούμενη διαφάνεια μας είχατε πει ότι τα έξυπνα δίκτυα έχουν αυξηθεί κατά 50% και τα ε, σχέδια διοξιδίου του άνθρακα 25% αυξηθεί. Εγώ είμαι καθηγήτρια πανεπιστημίου και μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά όταν βλέπω τέτοια στοιχεία. Νομίζω ότι εσκεμένα θέλετε να δώσετε μία εσφαλμένη εικόνα και το βλέπουμε αυτό από την επόμενη διαφάνεια που μας ενημερώνει ότι Έχουμε πολύ λίγα σχέδια ακόμη για τα έξυπνα δίκτυα και το διοξείδιο του άνθρακα. Τα περισσότερα σχέδια αφορούν τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο. Οπότε, ακόμη και αν έχουμε αύξηση 50%, δεν αρκεί. Γιατί από το 0 μέχρι το 1 πάλι είναι 100% αύξηση. Αλλά ε, στην πράξη δεν σημαίνει τίποτα αν έχουμε μόνο ένα σχέδιο, ή δύο ή τρία. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μου σχόλιο. Ότι θα πρέπει να αρχίσουμε σταδιακά να εξοβελίζουμε τα ορυκτά καύσιμα από το ενεργειακό μας μείγμα. Θα πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά, οπότε θα πρέπει να απεικονίζεται αυτό και στον κατάλογο των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος. Θέλουμε φιλοπεριβαλλοντική ενέργεια για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές, άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε τέτοιου είδους σχέδια. Πώς βλέπετε στο μέλλον το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρόλο που δεν είναι ε, θεσμικά πολύ ισχυρό, νομίζω ότι έχει νόημα να έχουμε έντονο διάλογο κατά την προετοιμασία των σχεδίων. Γιατί είναι σημαντικό τα σχέδια αυτά να είναι φιλόδοξα και να ανταποκρίνονται στις ε, απαιτήσει και τις δικές μας, αλλά κυρίως της κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ. Κύριος Κασάρες. Κύριε Αναπληρωτή Γενική Διευθυντά, εγώ θα διαβάσω την επιστολή ε, που έλαβε η ομάδα μου στις 3 Φεβρουαρίου από τον Επίτροπο Μιγέλα Αρίας Κανιέτε και που αναφέρει ότι είμαι έτοιμος να αναμίξω περισσότερο τον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει των διοργανικών μας συμφωνιών κατά την, επιλογή ε, των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος πριν την αποκριστάλλωση του καταλόγου των σχεδίων αυτών. Επίσης θέλω να έρθουν οι στενοποί στις υποδομές σε κάποιες ευρωπαϊκές περιφέρειες και για το ε, κατάλογο των σχεδίων και των αναδόχων που προτείνονται. Γι' αυτό θα ήθελα να έχω πιο τακτική συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Ήτρε σε βασικές περιφερειακές συνεδριάσεις, ιδιαίτερα στα πλαίσια των συνεδριάσεων του, της υπορικής ομάδας υψηλού επίπεδου ε, ειλικρινός δικό σας, Μιγέλ Αρίας Κανιέτε. Αυτές είναι οι υποσχέσεις του Επιτρόπου, όπως φαίνεται στην επιστολή. Αλλά φαίνεται ότι αθετήθηκαν αυτές οι υποσχέσεις, γιατί συνεχίζει να είναι αδιαφανής ο τρόπος εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και η απροθυμία της να εμπλέξει ενεργά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην όλη διαδικασία. Πάμε τώρα σε αυτό το τέταρτο κατάλογο. Ο προηγούμενος, ο τρίτος κατάλογος, περιείχε πολλά σχέδια υποδομών με ορυκτά καύσιμα που θα μπορούσε να μπλοκάρει την απαλλαγή από το διοξίδιο του άνθρακα. Τώρα μας υποβάλλεται ένα νέο κατάλογο, τον τέταρτο, που έχει περιορισμένο αριθμό σχεδίων για το ορυκτά καύσιμα και έχουν αλλάξει αναλογίες μεταξύ ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Αλλά ως προς τη χρηματοδότηση, πώς θα εξορροπήσετε αυτά τα σχέδια, τα ηλεκτρικά και το φυσικό αερίου στον κατάλογό σας. Τέλος, μας προβάλλατε ως επιτυχία και φαίνεται ότι ε, είναι επιτυχημένη αυτή η σύνδεση της Ιβηρικής Χερσονήσου με τη Γαλλία από το βασκονικό κόλπο. 2,8% είναι το σχέδιο ποσοστό εφαρμογής και μάλιστα θα ε, διπλασιαστεί το ε, σε σχέση με το 2005. Πώς όμως θα υλοποιήσετε το 12% μέχρι το 2020 και το 15% μέχρι το 2030 με βάση τους στόχους που έχουμε. Σας ευχαριστώ κύριος Πέτερσεν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσίασή σας. Ε. Προφανώς. Μια και πήραμε τα έγγραφα μόλις χθες το βράδυ δεν ε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, αλλά θα έχουμε χρόνο να σχολιάσουμε στο μέλλον πιο συγκεκριμένα. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι πρόκειται να το κάνουμε. Θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Ξεκινήσατε λοιπόν ε, με τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα αντιευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα, τα οποία είναι στην καρδιά της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Προφανώς, αυτό στέκει. Πολύ ορθό. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Ποια είναι η διαδικασία σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση των κριτηρίων αυτών. Το συζητήσαμε, συμφωνήσαμε από αυτόν στην ε, κανονισμό ΣΕΦ την ε, άνοιξη. Το θέμα είναι ότι αν αναθεωρήσουμε τις κατευθυντήρες αυτές θα υπάρχουν διαφορετικές γραμμές σε ό,τι αφορά τις, ε, τα αρκετά καύσιμα και τις ανανεώσιμες πηγές καυσίμων. Θα υπάρχει λοιπόν μια διαφορετική ισορροπία. Θα πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση. Ρωτώ λοιπόν, πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία και πώς θα επηρεάσει αυτό τον κατάλογο που συζητάμε σήμερα. Αναθεώρησε λοιπόν το καφεντήρι γραμμών. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Πείτε μας παραπάνω. Κατά δεύτερον, όλοι αναμένουμε με αγωνία τι θα μας παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από 100 ημέρες όταν θα ξεκινήσει να περνάει ο χρόνος. Ε, να δούμε ποιες ε, φιλοδοξίες θα έχει να επιδείξει στην ενέργεια και στην ενεργειακή πολιτική. Θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει περιβαλλοντικές μελέτε αντικτύπου για το χαρτοφυλάκιο αυτό. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτό το χαρτοφυλάκιο με τα τεράστια αυτά έργα θα συνάδει με τι περιβαλλοντικές φιλοδοξίε που έχουμε θέσει. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα υλοποιηθούν. Γιατί θεωρητικά. Αν ένα μεγάλο κομμάτι του χαρτοφυλακίου έχει να κάνει με το πετρέλαιο και με το αέριο, πέρα από τις ισορροπίες, τι θα γίνει. Σε 10-15 χρόνια θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου τα όσα συμφωνήσαμε σήμερα θα είναι αντίθετα με τις φιλοδοξίες μας. Αυτές οι δύο ερωτήσει λοιπόν είχα να σας απευθύνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριος Μπλος από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δούμε την τελευταία διαφάνεια, αν θα θέλετε. Καταρχάς, ε, το 2018 είπε η Διεθνής Υπηρεσία ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τίποτα το οποίο να εκπέμπει του άνθρακα. Και τώρα θέλουμε πολλά να δρομολογήσουμε σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτά τα προγράμματα για το αέριο, για παράδειγμα. Πώς το δικαιολογείτε, λοιπόν αυτό και ύστερα. Ή μας εξηγήσατε ότι ήδη υπάρχει μία μείωση των ε, έργων με φυσικό αέριο και είπατε ότι για τα ρεκτά καύσιμα και τα σχετικά έργα η αναλογία είναι 3 ε, προς 1, αλλά αν κατάλαβα σωστά είπατε ότι 1,5 δις πάνε στο αέριο και 1,5 δις σε έργα με άνθρακα. Άρα η η διαφάνεια αυτή είναι ακριβή ή μήπω είναι παραπλανητική σε ό,τι αφορά τον κανονισμό TNE που ζητά ουσιαστικά να αναφέρονται και να φυτώνονται τα πιο πολλά κονδύλια σε σχέδια κοινού ενδιαφέροντο με το ηλεκτρικό. Πώ συνδυάζονται όλα αυτά. Ο συνάδελφο επίση ανέφερε το εξή. Είπατε για τα τέσσερα κριτήρια τα αναφέρατε βιωσιμότητα ένα εξ αυτών, αλλά δεν βλέπουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τη διαδικασία για την ε, αναθεώρηση του κανονισμού TNE για τα ενεργειακά δίκτυα, τα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. Πείτε μας, ε, τι θα γίνει για όλο τον κύκλο των προϊόντων, πώς θα εφαρμοστεί η οδηγία. Θα υπάρξει κάποια μελέτη εφικτότητας, ε, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, θα λάβατε υπόψη τα θέματα ε, του τι συμβαίνει εκτός Ευρωπαϊκής ε, Ένωση, για τα θέματα τα περιβαλλοντικά. Και αυτή, η, αυτός ο κατάλογος για τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος πώς συνάδει με τους στόχους μας για την αλλαγή του κλίματος. Η τα επιστημονικά στοιχεία μας μιλάνε για μείωση 65% τουλάχιστον διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2030. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζουμε η νέα να προτείνει μείωση 55% τουλάχιστον. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα έργα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια έργα, προγράμματα με πολλά χρώματα στον κατάλογο. Ξέρω ότι, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων έργων στην Κροατία, δεν υπήρχαν ε, αρκετή διαβούλευση με τους ε, εμπλεκόμενου φορείς. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι με τον νέο κανονισμό ε, τέτοια έργα δεν θα καταλήγουν στον κατάλογο για τα PCI, τα σχέδια και ενδιαφέροντο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έβαλα χρονικό περιθώριο, είπε η είπε για να μην περιορίσω του συναδέλφου. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριε Μπόρχαρτ. έχουμε την μνήμα τη συμπερίληψη του νοτίου διαδρόμου στα δίκτυα, τα ενεργειακά. Οπότε πώς θα εξασφαλίσουμε διαφοροποίηση των πηγών μας μέσω και μακροπρόθεσμα. Και πιστεύετε ότι έχουμε αρκετά κονδύλια επαρκή για τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρασνοντέμψκι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον καθηγητή Μπόρχαρτ για την παρουσίαση που μας έκανε και ευχαριστώ που μας υπενθύμησε και τους στόχους των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος. Ένας από τους στόχους αυτούς είναι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Θα πρέπει επίσης να σας υπενθυμίσω ότι εδώ στην Επιτροπή μας ασχολούμαστε και με την βιομηχανία, την στρατηγική για τη βιομηχανία και τη δημιουργία υποδομών που είναι μια χρονοβόρος διαδικασία. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το φυσικό αέριο και τους διάφορους τομείς ε, που επηρεάζονται και επίσης το θέμα της εξάρτησης ε, από τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Και ο εξυγχρονισμός σε θέματα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ήδη λαμβάνει χώρα σε κάποιες ε, χώρες μέλη. Και πολλές φορές ε, προσπαθούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο, εγκαταλείποντας τα ορυκτά καύσιμα. Δυνάμει και το στόχο μας ε, για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σας ρωτήσω πώς θα εφαρμοστεί την επόμενη πενταετία όλα αυτά τα σχέδια προκειμένου να υλοποιηθούν οι νέες φιλοδοξίες και οι νέοι στόχοι μας για το περιβάλλον. γιατί μερικές φορές ε, στο παρελθόν δεν υλοποιήσαμε τους στόχους μας και δεν εφαρμόσαμε το πακέτο αυτό. Οπότε, ίσως ε, δεν εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό μας, που είναι πρωταρχικός μας στόχος. Δεν θα πρέπει να διακυβεύσουμε αυτό το στόχο της ασφάλειας του ενεργειακού ε, εφοδιασμού μας. Πώς βλέπετε λοιπόν παράλληλα αυτές τις δύο διαδικασίες στην νέα κοινοβουλευτική θητεία σε σχέση με, τους, με τις εργασίες που είχαν γίνει στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και τους στόχους που είχαμε θέσει τότε. Ευχαριστώ. Από την Κούβα τώρα. Η ε, Κονιλία Ένιστα, να σας πω, ένας τέτοιο κατάλογος με τόσο μεγάλη έκταση που έχει τόσο μεγάλη σημασία να το λαμβάνουμε τελευταία στιγμή χθε το βράδυ και να το διαβάσουμε γρήγορα γρήγορα για να πούμε ναι, σήμερα και να το περάσουμε γρήγορα γρήγορα ως πράξη καταξιοδότηση, αυτό το θεωρώ πάρα πολύ περίεργο και πραγματικά δεν δείχνει σεβασμό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό κατάλογο και το καθοριστικό για μα είναι, κοιτώντα το κατάλογο αυτό, ανταποκρίνεται στι ανάγκε που έχουμε μια τέτοια εποχή κατά πολέμηση τη αλλαγή του κλίματο, Όλα αυτά που μπαίνουν εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω με βάση ποια κριτήρια αναπτύχθηκαν όλα αυτά. Πώς τα έχετε φανταστεί. Για μένα αυτή η λίστα, αυτός ο κατάλογος είναι μια λίστα του τελευταίου αιώνα. Εμείς άλλα προγράμματα, άλλα έργα θέλουμε να ενισχύσουμε και να προωθήσουμε. Αυτά που μας ε, βρίσκει σύμφωνος είναι η ενίσχυση των ε, διασυνδέσεων. Ναι, αυτό μάλιστα. Αλλά σε ό,τι αφορά το αέριο, κοιτώντα ε, τι έχουμε εδώ, αυτούς τους αγωγούς, αυτούς τους διαδρόμους αερίου που θέλουμε να προκύψουν. Προ τα που επενδύουμε. Έχουμε 25 ΜΚΟ που έχουν στραφεί στην ε, Τράπεζα Επενδύσεων και είναι κατά των προγραμμάτων αυτών. Έχουμε ακτιβιστές οι οποίοι είναι στη φυλακή γιατί έχουν πολεμήσει τόσο πολύ κατά των προγραμμάτων αυτών. Εμείς τα υποστηρίζουμε λοιπόν. Η υποστήριξη των υποδομών αερίου έχει κοστίσει δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Εμεί το μειώσαμε κάπω το ποσό αυτό, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε ουσιαστικά. Δυσκολεύουμε, δυσκολεύουμε πάρα πολύ και χρειαζόμαστε πολύ πιο πολλέ επενδύσει σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Το οποίο είναι γελίο, γιατί εδώ αφήνουμε να περάσει ένα κατάλογο. Κάνουμε επενδύσει σε ό,τι να είναι, αλλά όχι σε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε, ανανεώσιμε ενέργειε. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε λοιπόν το κατάλογο αυτό και πραγματικά πιστεύω ότι είναι και να σα πω την αλήθεια το πώς ε, αντιμετωπίζετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα θα πρέπει να αρχίσω να επιβάλλω κάποια χρονικά όρια. Σας παρακαλώ λοιπόν να κάνετε ερωτήσεις μέσα σε ένα λεπτό. Ο κύριος Μπέρενσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή. Οι ενεργειακέ υποδομέ του μέλλοντο θα πρέπει να μα δίνουν όχι μόνο ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες που έχουμε για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Κοιτώντας λοιπόν τα ηλιακά πάρκα, χρειάζεται απαραίτητο, απαραίτητη ανάπτυξη για να μπορούν να έχουν αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, Ολλανδία, στο το Φρέιζε και Τρέντελ Έχουμε προβλήματα γιατί έχουμε φτάσει στη μέγιστη ικανότητά μας στον τομέα αυτό και αυτά τα προβλήματα θα παρουσιαστούν και σε άλλες χώρες τη στιγμή που θα αρχίσουν τα προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Θα ήθελα λοιπόν να το επισημάνω αυτό το θέμα. Και σε ό,τι αφορά τα διεστηνωριακά αυτά έργα. Ιδάλω, ε, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στι φιλοδοξίε μα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μετάβαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάιρ. Ευχαριστώ Ε, έγιναν πολλές κριτικές, ε, συμφωνώ και εγώ, για την ε, καθυστέρηση στην, σε ό,τι αφορά την παραλαβή της λίστας αυτής. Καταφέραμε να ρίξουμε μια ματιά, θα τα κοιτάξουμε και πιο ενδελεχώς όλα αυτά. Να πω όμως λίγα πράγματα σε ό,τι αφορά τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Όλοι περιμένουμε να γίνουν κάποια συγκεκριμένα βήματα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή τροφοδοσία. Κύριε Μπόιχερ, Πώς ε, θεωρείτε ότι ενδεχομένω να βρεθούμε σε μια κατάσταση carbon locking. Διαβάζουμε σε κάποια σημεία στα έγγραφα ότι τα θέματα των αγωγών, τα σχέδια αγωγών θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για υδρογόνο και για άλλα στοιχεία πέρα από το αέριο. Should be, λέει στα αγγλικά. Αυτό δεν είναι υποχρέωση, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό ισχύει για όλα τα έργα με αγωγούς. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μετατροπή για άλλα αέρια. Το θέμα των αγωγών τώρα επίσης συμφωνώ σε ό,τι αφορά τους συναντέλφου που έβαλαν ένα ερωτηματικό για το κατά πόσο χρειάζονται τέτοια αγωγή ακόμα σήμερα. Θα ήθελα να μου πείτε τι υποχρεώσεις έχουμε. Στη σελίδα 11 αναφέρεται ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Connecting Europe Facility, από το ΣΕΦΕ. Ωραία. Υπάρχουν όμως άλλοι, άλλα σημεία κεφάλαια του προπολογισμού που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπέκαλινεν. Yes. <clears throat> Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να επικεντρωθώ στο θέμα των αυτοκινήτων. Γνωρίζουμε ότι τα αυτοκίνητα εκπέμπουν ε, διοξιδίου του άνθρακα 60% ε, περισσότερο από ότι ε, ο άνθρακας. Και είπατε ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των αυτοκινήτων. Οπότε, πιστεύετε ότι στο μέλλον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους α, αγωγούς για την παραγωγή και βιοαερίου, για τη μεταφορά βιοαερίου. Είναι πολύ σημαντικό να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αν όμως χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερα το αυτοκίνητο, δεν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Αν τα αυτοκίνητά μας και είναι ορυκτά καύσιμα. Ευχαριστώ. Κύριος Κομπίλιος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εγώ να επενέσω, να εγκομιάσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της και να εκφράσω την απόλυτη συμφωνία μου για τη συνάφεια της ενέργειας με τις κλιματικές αλλαγές. Αλλά υπάρχει και το θέμα το γεωπολιτικό και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Όταν μιλούμε για τη διασύνδεση των χωρών μελών μέσω των αγωγών αερίου, θυμάστε τι είχε γίνει με την Ουκρανία όταν έκλεισε τις τρόφιγες η Ρωσία. Επίσης, μιλούμε για ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να έχουμε όμως περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, θα πρέπει να την παράγουμε και τοπικά. Προς το παρόν ε, δεν έχουμε άλλες επιλογές από το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Πάντως από τον κατάλογο σας βλέπω μια σαφή προτεραιότητα για την εξασφάλισε το, των δικτύων ηλεκτρισμού των τριών χωρών της Βαλτικής και χαίρομαι γιατί και εγώ από τη Λιθουανία κατάγομαι οπότε η ασφάλεια του εφοδιασμού μας είναι ιδιαίτερα προσφυλής. Οπότε είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διασύνδεσή μα με τι υπόλοιπε χώρε. Διατέλεσα και πρωθυπουργό τη πατρίδα μου και θα προτιμούσα να είναι ακόμη πιο ενισχυμένο ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη φάση τη εκτέλεση των σχεδίων αυτών, κατά τη φάση τη εφαρμογή του γιατί η εφαρμογή ενός σχεδίου εξαρτάται από τρεις ή τέσσερις χώρες. Είναι διασυνοριακά αυτά τα σχέδια. Οπότε σε μια περιφέρεια μερικές φορές είναι δύσκολο και μεταξύ μας να συμφωνήσουμε για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε και να επιτελείται σωστά το έργο. Οπότε η ερώτησή μου είναι ξεκάθαρη. Πώς βλέπετε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη φάση της εφαρμογής των σχεδίων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίστο. Δεν ζήτησα το λόγο. Αλλά μια και με πολιτικό θα... και μου απευθύνεται την έκκληση να λάβω το λόγο, θα ανταποκριθώ. Μιλήσατε για περιορισμό των επενδύσεων στο φυσικό αέριο, αλλά θα ήθελα να μου πείτε γιατί ποσό μιλούμε, γιατί ε, δεν αρκεί μόνο ο λόγος μεταξύ των διαφόρων σχεδίων. Δεν μας δίνει μια ιδέα για την κλίμακα των επενδύσεων. Επίσης, θέλουμε νέες υποδομές ώστε να απεγκλωβιστούμε από τις υποδομές ε, ορυκτών καυσίμων. Οπότε, πώς θα, πότε θα χρησιμοποιηθούν αυτή αυτοί οι νέοι αγωγοί. Θέλουμε ένα φιλοπεριβαλλοντικό αέριο και με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να εγκρίνουν τα σχέδια. Να χρησιμοποιούνται αυτή η αγωγή και για τη μεταφορά αερίου που θα είναι πράσινο, οικολογικό. Πώς θα εφαρμοστούν λοιπόν αυτά τα σχέδια. Επίσης, για τα σχέδια του φυσικού αερίου, η μείωση του, σχεδίου, του αριθμού των σχεδίων φυσικού αερίου οφείλεται στην, αυστηρότητα των της... στην αυστηρότερη επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στην έλλειψη σχεδίων από τα κράτη-μέλη ε, με θέμα το φυσικό αέριο. Ευχαριστώ. Κυρία Κουντάτσαρ, ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την παρουσίαση που μας έκανε και για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Όλοι εδώ συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε πιο καθαρές φιλοπεριβαλλοντικές μορφές ε, παραγωγής ενέργειας. Και αυτός είναι και σημαντικός ε, στόχος, από τους πιο σημαντικούς, του Μηχανισμού Συνδέοντας στην Ευρώπη, του ΣΕΦ. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι οι στόχοι αυτοί θα επισκιάσουν τις γεωγραφικές μας προτεραιότητες, γιατί έτσι θα υπονομεύσουμε το στόχο της καταπολέμησης της ενεργειακής απομόνωσης και την εξασφάλιση ισότιμων ευκαιριών σε όλου του καταναλωτές στην Ευρώπη, γιατί και αυτή είναι αξιοσημείωτη στόχη των νέων σχεδίων. Θα σας δώσω την το παράδειγμα της ε, πατρίδας μου, της Μάρτας, που ακόμη δεν είναι συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό, ε, αερίου. Αυτό οφείλεται στον ισιωτικό χαρακτήρα μας που μας κρατάει υπομονωμένους. Είναι σημαντικό να έχουμε διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, αλλά χρειαζόμαστε και τις απαραίτητες υποδομές σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως είπατε κι εσείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην αφήσουμε κανέναν πολύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πίσω. Επίσης, θέλουμε να στηρίξουμε τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος και ο μηχανισμός συνέντας στην Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προωθήσει τέτοια σχέδια και στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ κυρία Κουτατσάρ. Κυρία Κλόκ. Ε, κυρία Κλότς μάλλον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. η σαν πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στην επιστολή ανάθεση καθηκόντων ε, για την Επίτροπο Ενέργειας, ε, αναφέρεται στο σημαντικό ρόλο του φυσικού αερίου για τον περιορισμό των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα. Και μάλιστα στη διάρκεια της ακρόασης η οριστής Επίτροπος Σίμψον το επιβεβαίωσε ότι θα έχει σημαντικό μεταβατικό ρόλο το φυσικό αέριο. Τι θα πούμε όμως στην Συλλησία. Συμφωνώ με την κατάσταση αυτή, γιατί οι νέες οικολογικές πολιτικές ασκούν τεράστιες πιέσεις σε εθνικές οικονομίες όπως της Πολωνίας, που είναι εξαρτημένη από τον άνθρακα, αλλά και ε, στις οικονομίες άλλων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Είναι προφανές ότι το φυσικό αέριο είναι η μοναδική απάντηση και μοναδική λύση που θα έχουμε στο μέλλον. Αλλά εμείς, χώρες όπως η Πολωνία, δεν είμαστε έτοιμοι για τόσο ε, απότομο ε, εξυγχρονισμό, ούτε τόσο ε, μετάβαση σε νέα οικονομία. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποια ευαίσθητα στρώματα του πληθυσμού και κάποιες πιο ευάλωτες περιοχές. Γιατί ακούω ότι πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αλλά ο άνθρωπος ποια θέση έχει σε όλα αυτά. Το πιο σημαντικό δεν είναι το κλίμα, αλλά ο άνθρωπος. Γιατί αν δώσουμε μεγαλύτερη έφαση στο κλίμα από ό,τι στον άνθρωπο, είναι σαν να αρνούμαστε την σημασία που έχει ο άνθρωπος στον πλανήτη. Επίσης, ε, ε, πολλές ε, μεγάλες επιχειρήσεις ε, αποκομίζουν τεράστια κέρδη με την πολιτική αυτή και την πληρώνουν οι φτωχότεροι συμπολίτε μας. Αυτό είναι πραγματικά άδικο, αντικοινωνικό και αγνοεί και το θέμα της ε, ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Αν εμείς σταματήσουμε, ε, κλείσουμε τα θρακοριχεία μας ή στραφούμε μόνο στο φυσικό αέριο, τότε πραγματικά θα γίνουμε, θα εγκλωβιστούμε στην ρωσική ομπρέλα και θα διονυστεί αυτή η εξάρτησή μας από τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Μπόχβαντ. Στην παρουσίασή σας ε, μιλήσατε για τους τρεις πυλώνες ε, ε, διασφάλιση προμήθειας, αποδοτικότητα αν αυτό είναι αυτό που εννοείται Green Deal, ε, δεν φτάνει. Έχετε ε, φυσικά το πακέτο για τα ΕΦΗ e δίκτυα, αλλά υπάρχει πάντα το πρόβλημα ε, των ορυκτών καυσίμων. Στο Σάνον, ας πούμε, ανήκει στο 5-3 και θα πρέπει να εισάγουμε φυσικό αέριο βρώμικο που προέρχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείες το οποίο έχει ίχνος ε, διοξιδίου άνω του 40% από άλλα φυσικά αέρια. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν ποιος μπορεί να βγάλει το πρόγραμμα αυτό από τον κατάλογο. Η Ιρλανδία, το κράτος μέλος θα αποφασίσει ή αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απάντησή σας τι περιμένω με ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να μάθω αν έχετε κάνει μια αξιολόγηση του περιβαλλοντικού ίχνους των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Ο κύριος Κεράμ. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή για την παρουσίασή του. Δεν μπορούμε να στουρφοκαμιλίζουμε πλέον. Κάθε χρόνο τα στοιχεία είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Ήδη από το 2014, παρόλα αυτά από τότε έχουμε δώσει 1,5 δις σε ορυκτά καύσιμα ε, και συγκεκριμένα σε φυσικό αέριο. Δεν παίρνουμε μέτρα εναντίον της κλιματολογικής κρίσης και θα πρέπει να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε ε, προγράμματα τα οποία είναι ε, αντίθετα με την χάρτα των Παρισίων. Η γαλλική αντίστοιχη υπηρεσία χθες ε, δεν μπόρεσε να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Δεν μπορούμε εμείς να υιοθετούμε σε εισαγωγικά, το βάζουμε, κλιματοκτόνα μέτρα και δεν προστατεύουμε έτσι τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ακούσατε τις απόψεις των συναδέλφων, όλοι ανησυχούμε από τις κλιματολογικές αλλαγές. Πρέπει να διαγράψετε ε, τα προγράμματα που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, να μην κάνετε καν δεκτές τις λογικές 3 προς 1 ή 4 προς 1, δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε καν αυτό το 1. Και να αναθεωρήσετε επίσης τον κανονισμό του 2013 για, για τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με την Χάρτα των Παρισίων πλέον. Κυρία Πάουλους, δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία ήδη έχουν υποθεί, θα ήθελα ίσως να προσθέσω κάποια σημεία. Η διασφάλιση προμήθειας ενέργειας περιλαμβάνεται στους στόχους και από ό,τι καταλαβαίνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει την προμήθεια ενέργειας, την ασφάλεια της ενέργειας σαν ασφάλεια προμήθειας ενέργειας. Στη Γερμανία σαν παράδειγμα ε, ε, Κάποιες ε, μονάδες παραγωγής όταν έκανε πάρα πολύ ζέστη το καλοκαίρι του 18 δεν λειτουργήσαν σωστά γιατί δεν είχαν επαρκές ψυκτικό υλικό. Αλλάζουν λοιπόν τα πράγματα σε όλα τα επίπεδα. Πέραν τώρα των αριθμών τους οποίους μας δώσατε, υπάρχουν αρκετά προγράμματα τα οποία έχουν συν, συνενωθεί, έχουν συμπτυχθεί και το 5 προς 1 έγινε 6 προς 2 ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι τεχνητή η αλλαγή δηλαδή. Και τέλος να πω ότι το φυσικό αέριο δεν είναι χαμηλής απόδοσης σε διοξίδιο του άνθρακα. Γιατί αν δει κανείς ε, τις, ε, τα, τα ίχνη ε, του μεθανίου και της έκκλησης μεθανίου, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ότι με το διοξίδιο του άνθρακα. Να ακούσουμε τον κύριο Βέγκο για τι απαντήσει σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σα, για τι ερωτήσει σα. Δυστυχώ ε, στην παρούσα φάση δεν έχω τη δυνατότητα να απαντήσω σε όλε τι ερωτήσει μία προ μία. Νομίζω ότι θα ομαδοποιήσω κάποιε ερωτήσει και μετά θα αναφέρω και ενδεικτικά κάποιε άλλε. Καταρχά, αναφέρθηκε η κριτική ότι το στείλαμε το έγγραφο, το έγγραφο αυτό ε, πολύ αργά. Θα μπορούσαμε να έχουμε στείλει και τίποτα. Γιατί εμείς ολοκληρώσαμε την εργασία μας και το ερώτημα ήταν να το στείλουμε την προηγούμενη, το προηγούμενο βράδυ ή να μην το στείλουμε καθόλου. Ξέροντα ότι έχουμε τη σημερινή συζήτηση, ξέρουσαμε ότι θα ήταν ωφέλιμη μια αρχή τέτοια τη συζήτηση. Είναι μόνο η αρχή, δεν είναι το τέλος της συζήτησης. Δεύτερη παρατήρηση. Άκουσα πολλούς να λένε ότι τίθεται θέμα βιωσιμότητας, κάποιοι άλλοι να φωνάζουν ότι θα πρέπει να στραφούμε προς την ενεργειακό εφοδιασμό και την ασφάλεια εφοδιασμού. Εγώ δεν ε, το πιστεύω, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει και τους τρεις γενικούς ε, στόχους της ε, ενεργειακής πολιτικής βιωσιμότητα, ασφάλεια εφοδιασμού και εφικτότητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι απαραίτητα και προφανώς θα πρέπει να συνδυαστούν και φυσικά σε ό,τι αφορά και την ενεργειακή πολιτική δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Αυτή θα είναι η πρόκληση του μέλλοντος λοιπόν το πώς θα καταστήσουμε αυτό το τριπλό δίλημα αν θέλετε συμβατό. Πώς θα το κάνουμε να συνάδει με την Πράσινη Συμφωνία. Αυτή είναι η πρόκληση της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την οποία θα αναλάβουμε. Το μεγάλο τώρα θέμα στη συζήτησή μας, πολλοί το συζήτησαν και το έθιξαν, ότι είναι πάρα πολλά τα προγράμματα και τα έργα για το αερίο κτλ. Ε, να μην τα ξαναπώ. Αυτό που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω είναι το εξή, ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πώ έχει σήμερα η κατάσταση και πώ θέλουμε να είναι στο μέλλον η κατάσταση. Αυτό που συζητάμε στο α, τρέχον σχέδιο κοινού ενδιαφέροντο και στη λίστα είναι τι γίνεται τώρα. Γιατί τα πιο πολλά από τα προγράμματα για το αέριο ήταν στην λίστα αυτή από την πρώτη λίστα. Για τους λόγους που ανέφερε ο κύριος Κρασνοντεύσκη και ο κύριος Εκμπηλίους, για τους ίδιους λοιπόν λόγους, για ενεργειακή ασφάλεια, ασφάλεια εφοδιασμού. Μην ξεχνάμε ότι πριν από τρία-τέσσερα χρόνια έγινε μια τεράστια συζήτηση για την ε, κρίση του αερίου, την εξάρτηση από τις ρωσικές εισαγωγές και υπό την πρωτοβουλία για την Ενεργειακή Ένωση προτείναμε την διαφοροποίηση των υποδομών, των προμηθευτών και όλα αυτά μπήκαν στην πολιτική μας. Τώρα, τα έργα αερίου αποτελούν μία άμεση απάντηση για την πολιτική αυτή. Τώρα, επειδή αλλάζουμε την επικέντρωσή μας από την ενεργειακή ε, ασφάλεια, την ασφάλεια εφοδιασμού, τη βιωσιμότητα, θα πάνε χαμένα τα έργα αυτά. Δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Όπως είπε και η κυρία και αυτά είπε και η Ούρσουλα Φαντελάιεν, αυτό που είναι σαφές για μας είναι το εξή. Για το άμεσο μέλλον, για την επόμενη δεκαετία, θα εξακολουθήσουμε να χρειαζόμαστε το φυσικό αέριο. Θα πρέπει να επιτρέψουμε σε χώρες οι οποίες εξαρτώνται πολύ από τον ηλεκτρισμό από τον άνθρακα να έχουν την δυνατότητα να εγκαταλείψουν τον άνθρακα όλο και πιο γρήγορα, να τον αντικαταστήσουν με αέριο, γιατί οι χώρες αυτές δεν μπορούν στο χρονοδιάγραμμα που όλοι θέλουμε να εγκαταλείψουμε τον άνθρακα να εγγυηθούν ασφάλεια εφοδιασμού με ανανεώσιμες ενέργειες. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Δεν μπορούμε να παίρνουμε έργα τα οποία ήδη έχουν ε, μερικώς ε, χρηματοδοτηθεί και αναπτυχθεί και να τα βγάλουμε από τη λίστα και να πούμε «Α, κοιτάξτε, όλα αυτά ωραία ήταν μέχρι χθε, αλλά για αύριο θέλουμε κάτι άλλο». Έτσι έχει η κατάσταση. Εκεί που όλοι είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μεγαλύτερος προσανατολισμός για το κλίμα, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μέλλον. Και όντω οι τρει ε, γενικότεροι στόχοι θα πρέπει να συνάδουν με αυτό που ονομάζουμε Green Deal, Πράσινη Συμφωνία. Το ίδιο ισχύει και για τι υποδομέ. Πώ θα γίνουν αυτό, αυτά σε ό,τι αφορά τα θέματα ουσία και πώ θα τα πετύχουμε και με συγκεκριμένα κριτήρια. Επί τη ουσία είναι σαφέ ότι τα μελλοντικά έργα για το αέριο θα πρέπει να έχουν ε, πολλαπλές ε, λειτουργίες. Θα πρέπει τμήμα των προϋποθέσεων να σχετίζεται με τη δυνατότητα μεταφοράς πράσινων αερίων, υδρογόνου κτλ. Επίσης, ε, έχουμε και τους αγωγούς. Πώς όλα αυτά λοιπόν έχουν, συνδυάζονται με το υδρογόνο. Μπορούν να συνδυαστούν. Δυστυχώς όχι. Όχι όλα όχι όλη η αγωγή, γιατί μιλάμε για διαφορετική σύνδεση και για διαφορετική ε, διάβρωση όταν χρησιμοποιούνται οι αγωγοί για υδρογόνο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν το Connecting Europe Facility για την, ε, και τα σχετικά ενδιαφέροντος για να υπάρξει προσαρμογή των ε, αγωγών προκειμένου να υπάρχει την δυνατότητα μεταφοράς και πράσινων αερίων. Αυτό λοιπόν δεν αναφέρεται στο σημείο αυτό. Και αυτό γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η πιο αποφατική υποδομή είναι μια υποδομή η οποία θα μπορούσε να συνδυάσει το τα δίκτυο ηλεκτροδότησης με το δίκτυο αερίων. Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί τεχνικά, αλλά παίρνει χρόνο. Δεν θα το πετύχουμε αύριο. Πώς θα το πετύχουμε λοιπόν, αξιολογούμε στην ε, παρούσα φάση το κανονισμό για τα 10 χρόνια θα υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια συγκεκριμένη πρόταση με συγκεκριμένε προτάσεις μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους και αυτό αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά που συνόψισα ως άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα σε μεγαλύτερο βάθος και να συζητήσουμε τι γίνεται και με θέματα ε, μελέτης εφικτότητας και περιβαλλοντικής εφικτότητας και βιωσιμότητας. Αυτό δυστυχώ δεν το κάνουμε ακόμα και λείπει από τον κατάλογο των κριτηρίων μας. Θα πρέπει να προσταθεί, το ξέρει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιο το έφτιαξε και ζήτησε να πούμε τι γίνεται με τα έργα πετρελαίου. Προφανώ και αυτό δεν έχει θέση στη λίστα σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος. Είναι τμήμα του παρελθόντος. Τι να κάνουμε όμως που είναι τμήμα του κανονισμού δεκαετίας ε, κατά το παρελθόν είχε να κάνει με την ε, βιομηχανία δηληστηρίων. Ε, θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται και με κάποια ηλεκτρονικά καύσιμα και με άλλα καύσιμα τα οποία δεν παράγονται από πετρέλαιο. Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ε, Κάποιο είπε ε, κατά πόσον υπάρχει χρηματοδότηση από του ΕΦΕ. Νομίζω ότι όχι. Από όσο ξέρω δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα χρηματοδότηση από, ευρωπαϊκά, από ευρωπαϊκού πόρου. Ύστερα, ετέθησε το θέμα τη χρηματοδότηση εδώ. Για να αναφερθώ στην ε, κυρία Ερβάν. Το είπα και στα αριθμητικά στοιχεία. Αν έχουμε δύο έργα και προσθέσουμε άλλο ένα, τα ποσοστά είναι εκπληκτικά. Γι' αυτό και σας έδωσα τις αναλογίες και νομίζω ότι αυτό αποτελεί πιο ακριβή αποτύπωση της πραγματικότητας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε συγκεράσει έργα. Κάποιο ρώτησε κατά πόσον αφήσαμε κατά μέρο κάποια έργα. Όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ αυστηρή και καλά έκανε. Γιατί αγωνιστήκαμε να βγάλουμε κάποια έργα. Η κυρία Κουταγιά έθιξε ένα άλλο ε, έργο το οποίο αφαιρέσαμε η διασύνδεση μεταξύ Μάλτας ε, και Ιταλίας για το αέριο. Εδώ να σας πω ότι ίσως για πρώτη φορά τα κριτήρια βιωσιμότητας ε, τηρήθηκαν. Γιατί αφαιρέθηκε λοιπόν το σχέδιο αυτό, αυτό το έργο. Γιατί από πλευράς, από τη χρηματοδότηση είναι ακόμα στη λίστα ε, PCI σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος. Γιατί λοιπόν, γιατί στην πρόταση χρηματοδότησης δεν ήταν σαφές ποια θα είναι η μελλοντική στρατηγική της Μάλτας. Ε, επειδή έχετε ήδη γραμμή ηλεκτρικού με την Ιταλία, έχετε μια, ένα πλωτό ε, σταθμό και τώρα θέλετε και έναν αγωγό για αέριο με την Ιταλία. Το ποσοστό για τις ανανεώσιμες που αναφέρατε ήταν αρκετά μετριοπαθές. Όλα αυτά λοιπόν από κοινού μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούσαμε να προτείνουμε το έργο αυτό για χρηματοδότηση γιατί ήταν εντελώς ασαφές ποιες ήταν οι προθέσεις σας σε ό,τι αφορά αυτόν τον αγωγό. Γιατί εκεί είναι ο κίνδυνος. Αν σήμερα βάλουμε ένα τέτοιο αγωγό ε, στο νερό, θα μείνει εκεί τα επόμενα 50 χρόνια. Και γι' αυτό λοιπόν εξετάζουμε και τη μελλοντική διάσταση των έργων αυτών. Τι γίνεται στο μέλλον με τους αγωγούς αυτούς. Θα πρέπει να είναι αμα, αγωγή πολλαπλών χρήσεων. Αν θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Άλλα έργα τα οποία βγάλαμε από τη λίστα, γιατί θεωρούσαμε ότι δεν ήταν κατάλληλα. Πραγματικά λοιπόν εξετάσαμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πω καταρχάς ότι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασφαλώς στη διαδικασία αυτή που είναι πράξη κατά εξουσιοδότηση κατοχυρώνεται στη συνθήκη το δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει την τελική ε, εγκεκριμένη ε, πράξη κατά εξουσιοδότηση. Αλλά έχετε δίκιο. Και ο Επιτροπός, ο κ. Κανιέτε, έχει την αίσθηση και εμείς ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί στην ανάπτυξη και την κατάρτιση της λίστας και μάλιστα σε πρώιμο στάδιο. Γι' αυτό α, ανοίξαμε την περιφερειακή ομάδα για τη συμμετοχή μελών του Κοινοβουλίου, βοηθών, εκπροσώπων, εν πάση περιπτώσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν ανοιχτή η διαδικασία αυτή και κάποιοι συμμετείχαν, άλλοι δεν συμμετείχαν. Ίσως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία αυτή, αλλά σε όλη την διαδικασία αυτή. Όποτε έγιναν εργαστήρια, όποτε έγιναν συναντήσεις, ήταν ανοιχτά και είχαν αποσταλεί και προσκλήσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Και όπως σας είπα, γιατί μας είπατε ότι δεν είναι διαφανή η διαδικασία, όλες αυτές οι συναντήσεις ήταν επίσης μεταδιδόμενες στο διαδικτύο. Επίσης, μία άλλη ερώτηση. Για την... το στόχο διασυνδεσιμότητας μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας 2,8 είπατε, σωστά. όντω δεν μα ικανοποιεί αυτό το ποσοστό, είναι χαμηλό. Έχουμε πολλά κονδύλια ε, του μηχανισμού συνδέοντα στην Ευρώπη ε, στο βασκονικό κόλπο. Και αυτό είναι από τα πιο σημαντικά σχέδια ε, για τα υποβρύχια καλώδια. Και παρόλο που έχει διπλασιαστεί το ποσοστό, εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Αυτό ισχύει για πολλού και διάφορους λόγους. Ο ένας είναι η αντίσταση της κοινωνίας, η αντίσταση των πολιτών. Ε, δεν θέλουν να, να έχουμε πολλά καλώδια πάνω από τα πυρηναία. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε σοβαρά, γιατί θα μας ε, προβληματίσει και στις μελλοντικές μας υποδομές. Οι ανάδοχοι των έργων θα πρέπει να εμπλέκουν την κοινωνία των πολιτών σε πρώιμη φάση, να εξηγούν ε, τις προθέσεις τους ε, έγκαιρα και όχι όταν ε, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας ε, ήδη ζητούν άδεια για την εκτέλεσή του. Τι άλλο μου έμεινε. Ελπίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα τουλάχιστον σημεία. Α, και το θέμα του Σάνων. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα ε, και μας διαφωτίζει για τα προβλήματα που έχουμε σήμερα και εμείς. Τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος βρίσκονται στα χέρια των κρατών μελών, γιατί είναι προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και μετά πηγαίνει στις περιφερειακές ομάδες. Εμείς, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν λαμβάνουμε τις προτάσεις, θα πρέπει, πρέπει να ακολουθούμε σαφείς κανόνες. Δεν μπορούμε να κρατάμε ένα σχέδιο στον κατάλογο αν ένα κράτος μέλος είναι κατά. Και εν προκειμένου αυτό ίσχυσε. Απ' την άλλη πλευρά, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και γίνει και ανάλυση κόστους-οφέλους που δείχνει θετικό λόγο κοινωνικής ευημερίας, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να το συμπεριλάβουμε στον κατάλογο. Και όπως επισήμανε και ο κύριος Πίτερσον, και το δέχομαι, εδώ υπάρχει ένας χαμένος κρίκος στο σύστημα που θα πρέπει να τον προσθέσουμε στο, στα μελλοντικά σχέδια. Θα πρέπει να έχουμε έναν ουσιαστικό έλεγχο, μια ε, πραγματική αξιολόγηση της συμβατότητας του σχεδίου με την κλιματική μας πολιτική. Και σας έδωσα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ένας αγωγό φυσικού αερίου δεν θα πρέπει μόνο φυσικό αέριο να μεταφέρει. Θα πρέπει να είναι πολλαπλών χρήσεων, πολυλειτουργικό. να μπορεί να μεταφέρει και άλλα και άλλες ουσίε θα ενισχύσουμε τον ψηφιακό εμπλουτισμό των έξυπνων δικτύων. Όλα αυτά θα μας ε, οδηγήσουν σε καλύτερη αντίληψη της κατάστασης. Και τέλος, γιατί αναφέρθηκε το τερματικό υγροποιημένο φυσικό αερίο στο ΚΡΚ της Κροατίας και τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων. Όντως, στο ΚΡΚ είχαμε αυτό το πρόβλημα στην Κροατία με το τερματικό LNG. Και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνάδελφοι από τη Γενική μου Διεύθυνση, έστειλαν στους Δήμους πρόσκληση για διαβουλεύσεις. Γιατί υπήρχε ένα εσωτερικό πρόβλημα και προσπαθήσαμε να το λύσουμε πηγαίνοντας εμείς οι ίδιοι επί τόπου και ζητώντας απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και των Δήμων για, ζητώντας τη γνώμη τους για το τερματικό υγροποιημένο φυσικό αερίο στο ΚΕΡΚ. Εδώ δεν αφισβητείται η ίδια ιδέα του τερματικού, γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της υποδομής που χρειάζεται η ευρύτερη περιοχή, αλλά ο τρόπος και η λυπή συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών ε, ήταν ε, προβληματικός, γιατί δεν έγιναν έγκαιρες διαβουλεύσεις με τους ε, ενδιαφερόμενους. Θέλουμε λοιπόν στο μέλλον να εξασφαλίσουμε σε πιο πρώιμη φάση και πολύ πιο έγκαιρα τη συμμετοχή τη Συμφωνία των Πολιτών. Ευχαριστώ. Πάντω χαίρομαι γιατί κλείσατε με μια πολύ καλή ιδέα και μια δέσμευση για να εμπλέξετε σε πολύ πρώιμο στάδιο του εμπλεκόμενου φορεί και την κοινωνία των πολιτών σε τέτοιου είδου σχέδια. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρουσία σα, ευχαριστώ και του συναδέλφου για το ενδιαφέρον του. Όπω είπε και ο Γενικό Διευθυντή, βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας, οπότε είναι σημαντικό να αφογκραζόμαστε και τους ενδιαφερόμενους, ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Μπόκαρτ και σας περιμένουμε και στο μέλλον για τη συνέχεια της συζήτησης. So, dear if you can... Uh, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συνεχίσουμε. Καθίστε παρακαλώ. Κυρία Πάουλος και εσείς καθίστε. Για να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικείμενη Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών. Είναι μαζί μας σήμερα ο κύριος Ανδρέας Γκάης, που είναι τιματάρχης ε, του της πολιτικής ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον καλέσαμε για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων εν ώψη της Παγκόσμιας Διάσκεψης ραδιοπικοινωνιών που θα λάβει χώρα στο Σάρμελ Σέικ της Αιγύπτου 28 Οκτωβρίου με 22 Νοεμβρίου. Σχεδόν ένα μήνα θα κρατήσει. Φαντάζομαι σας ενδιαφέρει ο αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτή η παγκόσμια διάσκεψη ραδιοπικοινωνιών στην πολιτική ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, του φάσματος ε, για την τεχνολογία 5G, καθώς και την, ε, σε επιπτώσει που μπορεί να έχει στην διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Γκάι, έχετε το λόγο και θα ακολουθεί η συζήτηση με του συναδέλφου. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σας. Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαστε στο μετέχνιο. Θα σας κάνω μια ενημέρωση και θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Θα πω λίγα λόγια για τη διαδικασία, το περιεχόμενο και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, στις παγκόσμιες διασκέψεις ραδιοεπικοινωνιών. Η ITU είναι η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών και είναι ένας ε, ειδικό ε, οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιεί τις παγκόσμιες διασκέψεις ραδιοεπικοινωνιών. Συγκεντρώνει περίπου 3.000 εκπροσώπους από 193 μέλη του ΟΗΕ. Τώρα θα διαρωτάστε γιατί 3.000 άνθρωποι θέλουν να συζητήσουν τόσο λεπτομεριακά θέματα όπως είναι αυτό του ραδιοφάσματος και ε, άλλων περίπλοκων θεμάτων. Το κοινό αυτών των ε, συμμετεχόντων παρά την διαφορετικότητά τους είναι το εξής. Γιατί έχουμε και κράτη-μέλη στη διάσκεψη αυτή, αλλά και ε, χειρίστες ή παρόχους δορυφορικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, ε, κάποιες εφαρμογές στρατιωτικές, ραδιοστρονομία και όλοι αυτοί οι φορείς χρειάζονται το ραδιοφάσμα, χρειάζονται το φάσμα και θέλουν να το χρησιμοποιούν χωρίς παρεμβολές με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Είναι πολλοί λοιπόν οι φορείς που συμμετέχουν σε τέτοιες παγκόσμιες διασκέψεις ραδιοπικοινωνιών. Σκοπός αυτών των διασκέψεων είναι η επικαιροποίηση των κανονισμών ραδιοπικοινωνιών. Οι κανονισμοί ραδιοπικοινωνιών είναι συνθήκες που ρυθμίζουν τα διασυνοριακά θέματα της χρήσης φάσματος, γιατί το φάσμα δεν γνωρίζει σύνορα. Μεταδίδεται σε μεγάλες αποστάσεις. Ως εκ τούτου ε, αν δεν υπάρχει συντονισμός μπορεί να έχουμε επιζήμιες παρεμβολές. Η Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών λαμβάνει χώρα κάθε τέσσερα χρόνια περίπου και ουσιαστικά είναι το επιστέγασμα μιας χρονοβόρας και έντονης προπαρασκευαστικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η προηγούμενη Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών είχε γίνει το 2015 και αμέσως μετά ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την επόμενη, τη φετινή Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοπικοινωνιών. Και δεν εννοώ μόνο ότι συμμετείχα στην προετοιμασία τα κράτη-μέλη, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, γιατί είναι πολλοί οι ενεχόμενοι που λαμβάνουν από την αρχή μέρος της προετοιμασίας. Η Παγκόσμια Διάσκεψη ραδιοπικοινωνιών δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, δεν γίνονται ε, ομιλίες πολιτικού χαρακτήρα, ούτε ακολουθείται κανένα σημαντικό πρωτόκολλο, ούτε είναι κατά ανάγκη ψηλόβαθμοι ε, οι συμμετέχοντες, αλλά εξετάζονται κάποιες τροπολογίες στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών. Τι σημαίνει αυτό. Σας έχω παρουσιάσει εδώ ένα πίνακα με τρεις στήλες. Αυτές οι τρεις στήλες εκπροσωπούν τι διάφορε περιοχέ του κόσμου. Η πρώτη στήλη, η πρώτη περιοχή αφορά την Ευρώπη και την Αφρική, η δεύτερη περιοχή είναι η Βόρεια και Νότια Αμερική και η τρίτη περιοχή είναι η ε, περιοχή Ασίας και Ειρηνικού. Έτσι δημιουργείται ένα πλαίσιο για τους κανονισμούς ραδιοπικοινωνιών και έχουμε και υποσημειώματα που ε, υπησέρχονται σε τεχνικές λεπτομέρειες για την αποφυγή των παρεμβολών. Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία τώρα και τη διαδικασία. Πώς ε, γίνονται αυτά. Τα μέλη της Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, ε, κυβερνήσεις και ενεχόμενοι, εκπονούν μελέτες που ξεκινούν ήδη αμέσω μετά το πέρας της προηγούμενης παγκόσμιας διάσκεψης ραδιοπικοινωνιών. Ουσιαστικά λοιπόν πραγματοποιούν μελέτες και καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα που ουσιαστικά είναι προτιμόμενες ε, εκβάσεις ή προτιμόμενα αποτελέσματα που τις υποβάλλουν σε μια περίπλοκη και τεχνική έκθεση προπαρασκευαστική, το CPM Report, και χάρη στην έκθεση αυτή οι διάφορες πλευρές ε, αποκομίζουν καλύτερη, πιο ξεκαθαρή ιδέα για τις απόψεις των υπόλοιπων μερών και έτσι βρίσκουν μεθόδους για να διεκπαιρεώσουν καλύτερα τα διάφορα τμήματα τη ημερήσια διάταξη τη επόμενη παγκόσμια διάσκεψη, γιατί γνωρίζουν ποιε χώρες ε, ε, προτιμούν ποιε μεθόδους. Αυτή είναι η προετοιμασία σε επίπεδο Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, αλλά έχουμε και προετοιμασία ε, στην Ευρώπη. Η προετοιμασία αυτή γίνεται κυρίως μέσω της CEPT, της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ταχυδρομικών Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών, στην οποία συμμετέχουν ε, φυσικά ε, οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συνολικά 48 χώρες, ε, η Ρωσία, η Τουρκία και γενικώ χώρες της Ευρωπαϊκής Επίρου. Συμμετέχουν λοιπόν οι χώρες αυτές σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη και ε, με τη συγκέντρωση αυτών των απόψεων καταλήγουμε σε μια κοινή θέση που δεν την υπογράφουν κατά ανάγκη και οι 48 χώρε, μπορεί λιγότερε να την υπογράψουν. Οπότε και στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών μπορεί να έχουμε διάσταση απόψεων ή να υπάρχουν μερικέ κοινέ θέσει, αλλά όχι συνενετικέ κατά ανάγκη. Στη συνέχεια αυτές οι πληροφορίες ε, υποβάλλονται για συζήτηση στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Τώρα, ποιο είναι ο ρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλήρε μέλο, τακτικό μέλο τη Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να ε, υποβάλει προτάσει να κάνει διαπραγματεύσει. ή δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Αυτά είναι δικαιώματα των μεμονωμένων χωρών μελών. Από την άλλη πλευρά, έχουμε κάποιους συγκεκριμένους τομεί όπου κάποιες αλλαγές που γίνονται στους κανονισμούς των ραδιοεπικοινωνιών που έχουν δύναμη συνθήκης μπορούν να επηρεάσουν το ενωσιακό δίκαιο. Και σε τέτοιες περιπτώσεις η συνθήκη προβλέπει το άρθρο 218 παράγραφος 9 για παράδειγμα που προβλέπει ότι όλα τα κράτη-μέλη διαπραγματεύονται από κοινού ως ένωση βάσει της δεσμευτικής απόφασης που είναι απόφαση του Συμβουλίου και που ελήφθη εν ώψη αυτής της παγκόσμιας διάσκεψης ραδιο, ραδιοεπικοινωνιών. Και είναι δεσμευτική, επαναλαμβάνω, υποχρεωτική. Τι γίνεται σε περίπτωση διάσταση απόψεω στο CPT. Εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνουμε ως ενοποιημένο κοινό μέτωπο στην παγκόσμια διάσκεψη, για να μην αποδυναμώσουμε τη διαπραγματευτική μα θέση. Οπότε, ποιες είναι αυτές οι θέσεις που διαμορφώνονται. Οι θέσεις αφορούν πολλά και διάφορα θέματα. Εδώ έχουμε μόνο μία υπομάδα, υποκατηγορία των θεμάτων που μπορούν να συζητηθούν στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοπικοινωνιών. Αυτά τα θέματα μπορούν να επηρεάσουν το ενωσιακό δίκαιο. Είναι θέματα ναυτιλιακά, ασφάλεια και διαχείριση της κυκλοφορίας, αεροναυπηγικά, και εκεί το θέμα της ασφάλειας ε, στην αεροπλοή είναι σημαντικό. έξι στήματα μεταφορών επίσης ε, είναι αντικείμενο συζήτησης. Άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι οι διεθνείς ε, κινητές τηλεπικοινωνίες, 3G, 4G, 5G, οι συζητήσεις που περιμένετε για το 5G. Επίσης έχουμε τα Wi-Fi, τα τοπικά δίκτυα τα σύρματα και εκεί ε, εξετάζεται το επιπλέον φάσμα. Ε, κινητά συστήματα δορυφορικά σε συγκεκριμένη ε, ζώνη. Η, η μελλοντική, το μελλοντικό θεματολόγιο για την επόμενη ε, παγκόσμια διάσκεψη ραδιοπικοινωνιών που θα γίνει το 2023, που συζητάται όμως από φέτος ήδη ο προσδιορισμός αυτού του προγράμματος εργασιών του, της διάταξης. Θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές θέσεις ε, να συνάδουν με τις αντίστοιχες ε, κοινέ ευρωπαϊκές θέσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών. Τι κάνουν και τι δεν κάνουν τώρα οι κανονισμοί ραδιοπικοινωνιών. Είναι υψηλού επίπεδου καταρχήν και προσδιορίζουν ένα πλαίσιο για την κατανομή των συχνοτήτων προκειμένου να αντιμετωπίζονται διασυνοριακά θέματα όπως είναι οι επιζήμιες παρεμβολές. Οι κανονισμοί ραδιοπικοινωνιών συνήθως εγκρίνονται συνενετικά και μάλιστα τα κράτη-μέλη έχουν χρονοβόρες συζητήσεις ε, και προσπαθούν να διευκολύνουν συνένεση μερικές φορές με υποσημειώσεις γιατί ζητούμενο είναι η συνένεση για τα θέματα αυτά τη τροποποίηση των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών. Επίσης, διευκολύνουν κάποιε οικονομίες κλίμακος οι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών, αλλά δεν θέτουν προδιαγραφές ή πρότυπα για εξοπλισμό, ούτε προσδιορίζουν την ακριβή χρήση ή τη λεπτομεριακή χρήση. Αυτό γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Οπότε ακόμη και μετά τη λήψη αποφάσεων για την επικαιροποίηση του κανονισμού ραδιο, ε, ραδιοεπικοινωνιών χρειάζεται περαιτέρω μία ε, νοσιακή εναρμόνιση για να ξέρουμε ε, ποιες ζώνες θα χρησιμοποιούνται για το 5G, ε, τι, θα χρησιμο τι ζώνες θα χρησιμοποιούνται για το Wi-Fi, για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Αυτά είναι λεπτομεριακά ζητήματα που δεν προσδιορίζονται σε επίπεδο Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Και τελευταία διαφάνεια, τι με έλεγενέστε μετά την παγκόσμια διάσκεψη του 2019. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει την έκβαση της διάσκεψης, θα εκπονήσει μια έκθεση σχετικά και θα υποβάλει και προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της ε, διάσκεψης του 2019 ξεκινάει ο κύκλος προετοιμασίας για την επόμενη παγκόσμια διάσκεψη που έχει προγραμματιστεί για το 2023. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Θα σταματήσω εδώ και είμαι πρόθυμος να απαντήσω στις απορίες σας και να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Καβάλιο. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να υπογραμμίσω τη μεγάλη σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο συγκεκριμένο χώρο. Μπορείτε να είμαστε κάπως πιο συγκεκριμένοι για τις πιθανές επιπτώσεις σχετικά με την ε, ανάπτυξη του 5G κατά πόσον θα επηρεάσει το πρόγραμμα αυτό και πώς ακριβώς θα υπάρξει η συγκατοίκηση σε εισαγωγικά με τρίτες χώρες. και Πέρες. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας σχετικά με το 5G. ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει διάθεση από 3,7 με 3,8 GHz για βιομηχανική χρήση. Για τις ενδιαφερόμενες βιομηχανικές δραστηριότητες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λόγω της σημασίας του 5G λοιπόν, γύρω από το φάσμα 4, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει την ε, δυνατότητα ε, καθορισμού ενός εύρους φάσματος όπως το κάνει η Γερμανία. Äh, äh, Σχετικά με το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, σχολιάσατε τις διαφορές που υπάρχουν σε διαμεθοριακές χρήσεις. Αν υπάρχει δυνατότητα χρήσης του ιδίου φάσματος και συχνότητας για διαφορετικούς χρήστες ε, μέχρι τα 80 MHz, γιατί πάνω από αυτό τότε η εμβέλεια είναι πολύ περιορισμένη και γι' αυτό ακριβώς είναι χρήσιμο να συζητιούνται σε ένα διεθνές φόρουμ. Είναι σημαντικά αυτά που είπατε και για τις ε, κινητές μορφές επικοινωνίας. Δεν θέλει να χρησιμοποιεί κανείς το κινητό τηλέφωνο μόνο στη Γερμανία, πρέπει να μπορεί να το χρησιμοποιεί και στην Ιαπωνία. Πρέπει να συμφωνήσουμε και υπάρχει επίσης ε, και η χρήση από τις θαλάσσιες μεταφορές Διαφορετικές χρήσεις λοιπόν των διαφορετικών συχνοτήτων μετά πάνω από το 80 MHz είναι κάτι το οποίο δεν μου λέει τίποτα. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κύριε Γκάις, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση σχετικά με τις επιπτώσεις σε σχέση με την ανάπτυξη του 5G. Όπως είπα εξ αρχής, η ημερήσια διάταξη είναι καθορισμένη. Ξέρουμε ακριβώς τι θα συζητηθεί στα πλαίσια του 5G. Αυτή τη στιγμή τα εύρη συχνοτήτων τα οποία είναι υπό εξέταση έχουν προκαθοριστεί είτε για το 5G είτε τα λεγόμενα IMT. είναι εύρη συχνοτήτων ιδιαίτερα υψηλά στα πλαίσια του ε, φάσματος συχνοτήτων σε επίπεδο μιλιμέτρα από 44 GHz και πάνω. Και αυτό το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει διάσκεψη είναι να συμφωνήσει ποια εύρη συχνοτήτων θα χρησιμοποιηθούν για το 5G στο μέλλον. Αυτό δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο επηρεάζει τα ισχύοντα ε, για χαμηλότερα εύρη και για τα 2G, 3G και 4G. Αλλά πρόκειται για νέα εύρη τα οποία παρέχουν τα χαρακτηριστικά παροχής υψηλών ταχυτήτων gigabit λόγω των υψηλών συχνοτήτων όπως είπαμε. Συνεπώς θα εξετάσουμε συγκεκριμένα εύρη και ένα από τα δύσκολα θέματα της συζήτησης που θα γίνει είναι ότι η διάθεση συχνοτήτων για το 5G σημαίνει ότι κάποιες άλλες υπηρεσίες θα επηρεαστούν αρνητικά. Ε, αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν χρησιμοποιείται ήδη ένα εύρος. Όταν συζητάμε λοιπόν για τις τεχνικές προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ε, το, ο εξοπλισμός του 5G θα πρέπει να είναι συμβατός. Αυτό σημαίνει υψηλό ή χαμηλότερο κόστος ε, για τον παραγωγό του εξοπλισμού. Η μεγαλύτερη προστασία η οποία παρέχεται στις υπόλοιπες υπηρεσίες τόσο αυξάνει περισσότερο το κόστος του εξοπλισμού. Από την άλλη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να εξισορροπούμε αυτό που κάνουμε με το 5G με άλλες υπηρεσίες που επηρεάζονται. 26 ε, GHz που είναι σημαντικό ε, εύρος για το 5G. Κάτω από αυτό χρησιμοποιείται για γεωδεσικές μελέτες και για το Κοπέρνικους και δορυφορικές επικοινωνίες. Συνεπώς θα πρέπει να βρούμε λοιπόν τη σωστή ισορροπία προστασίας ανάμεσα στις διαφορετικές υπηρεσίες από τη μία ε, τις δραστηριότητες τις επιχειρηματικές την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί τα όρια αυτά έχουν σχέση με την προστασία των δορυφορικών επικοινωνιών όπως μέσω του Κοπέρνικους, όπως και η παρατήρηση της επιφάνειας της γης χωρίς παρεμποδίσεις και χωρίς αρνητικούς επηρεασμούς της ακρίβειας των δορυφορικών μετρήσεων. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει μια σαφής πολιτική ε, πλευρά που θα ληφθεί υπόψη. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το συγκεκριμένο εύρος που χρησιμοποιεί ήδη η Γερμανία για τις βιομηχανικές χρήσεις του 5G ε, 3,7 με 3,8 GHz. Η διάσκεψη δεν συζητά στοιχεία σε τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειας σε σχέση με την απόδοση εύρους είναι καρμοδιότητα των κρατών μελών να το κάνουν. Είχαμε μακρές συζητήσεις στο παρελθόν όταν υπήρχε η συμφωνία για τον κώδικα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ο ρόλος των μεμονωμένων κρατών. Και τελικά τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα διαθέσουν το συγκεκριμένο ευρώ. Αν η Γερμανία λοιπόν θέλει να δώσει το 3,7 με 3,8 αποκλειστικά για τις βιομηχανικές χρήσεις, αυτό είναι μια εθνική απόφαση. Και δεν πρόκειται εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναμειχθούμε ή να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Παρ' όλα αυτά συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη και παίρνουμε τα στοιχεία αυτά, να δούμε σε ποιο βαθμό επηρεάζεται και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και πού μπορούμε να κάνουμε οικονομίες κλίμακας. Αν προκρατήσει κανείς ένα εύρος για ένα συγκεκριμένο χρήστη, αυτό σημαίνει υψηλότερες, υψηλότερες τιμές στους διαγωνισμούς για άλλους χρήστες και αυτό έχει συμβεί στη Γερμανία. Η τελευταία ερώτηση είναι οι λεγόμενες παρε... Ε, παρεμβολές. Όταν οι παρεμβολές ε, είναι μέχρι τα 80 MHz, τι συμβαίνει, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα, τόσο μικρότερη είναι η απόσταση την οποία διανύουν τα ραδιοκύματα. Ένας αναμεταδότης κοντά στα σύνορα σαν παράδειγμα θα επηρεάσει μόνο μία μικρή περιοχή μεθοριακή όσο πιο ψηλά εκπέμπει. Αλλά ακόμα και σε εύρος φάσματος στα 800 ή 700 MHz τα οποία έχουμε συζητήσει για τις πιθανές παρεμβολές εκπομπέων και κινητών δικτύων, τότε οι αποστάσεις μπορεί να φτάσουν τα 150 χιλιόμετρα. Υπάρχει δηλαδή μια ουσιαστικά μεγάλη περιοχή που επηρεάζεται αρνητικά και θα πρέπει να μην αγνοούμε ότι κάποια από τα αιτήματα αυτά δεν είναι μόνο εδαφικά. Οι παρεμβολές μπορεί να επηρεάζουν την επικοινωνία εδάφους αέρος και υπάρχουν δορυφορικά συστήματα τα οποία εργάζονται σε εύρη συχνοτήτων πολύ υψηλότερα. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αναχώρα γιατί οι δορυφόροι έχουν ένα ίχνος το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο, μερικές φορές έχει υπηρετικό εύρος ή και μεγαλύτερο ακόμα. Συνεπώς λοιπόν ό,τι κάνει κανείς σε εδαφικό επίπεδο αυτό μπορεί να επηρεάζει τον δορυφόρο γιατί ο δορυφόρος είναι πολύ ευαίσθητος σε άλλου είδους τηλεπικοινωνίες και <clears throat> σε τέτοιες καταστάσεις <clears throat> έχουμε χαρακτηρίσει κατά αποκλειστικότητα προσβάσιμες ε, ορισμένες περιοχές ε, και ορισμένα τμήματα του φάσματος για κινητές ε, τηλεπικοινωνίες ή για κάποιο άλλο τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάφορα, τίποτα στα διάφορα, συνάδελφοι, αν όχι, η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 11 και 12 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ.